Okay, well, welcome everybody. Um, I have... Καλώς ήρθατε όλοι. Things I have to say before we get... Θα ήθελα να πω κάποια πράγματα πρωτού ξεκινήσουμε. Πρώτα απ' όλα, για τους τύπους υποθέτω, προτείνω να εγκρίνουμε το σχέδιο ημερήσιας διάταξης, δεν υπάρχουν ενστάσεις, θεωρείται εγκεκριμένοι. Τις ανακοινώσει θα τις κάνω στο τέλο, για προφανείς λόγους, διότι πρέπει να προχωρήσουμε στις βασικές εργασίες με τους υπουργού. Καλώς ορίζουμε τους υπουργούς ε, οικονομικών της Γαλλίας και της Γερμανίας. Ήδη έγινε με την Ουγγαρία, το Βέλγιο και την Ισπανία ο προγραμματισμένος οικονομικός διάλογο και το νέο μέσο για την ενίσχυση του δημοκρατικού διαλόγου για την οικονομική διακυβέρνηση σε επίπεδο ευρωπαϊκή Ένωση. βαίνει αισίω Περιμένουμε ακόμη τον πρόεδρο του Eurogroup στην Επιτροπή ΕΚΟΝ και πρόσφατα έμαθα ότι ο Υπουργό Οικονομικών τη Ιταλία θα έρθει στι 21 Ιανουαρίου στην Επιτροπή μα για το χρονοδιάγραμμα, για τις ερωταπαντήσεις. Οι πολιτικές ομάδες έχουν δώσει ήδη τα ονόματα των όσων θα χρησιμοποιήσουν το χρόνο ομιλίας. Έχουμε 14 ομιλητές. Αν έχουμε χρόνο περίσσιο στη διάθεσή μας δεν νομίζω. Το αντίθετο μάλλον θα περικόψουμε κάποιους. Έχουμε στον κατάλογο τους συντονιστές ή τους αναπληρωτές και άλλα μέλη της Επιτροπής σε βάση του κανόνα Ντεχόντ. θα ήθελα να σε υπενθυμίσω ότι εσχάτως υπεκύρωσαν αυτό οι συντονιστές, δηλαδή θέλουν χρονοθυρίδα πεντάλεπτη για τις ερωταπαντήσεις αν Εάν λοιπόν ε, ε, δαπανίσετε τα πέντε σα λεπτά για την ερώτηση, δεν θα έχετε απάντηση. Λοιπόν, στο 1,5 λεπτό θα χτυπάω το σφυράκι για να μην χρειαστεί να σα διακόπτω και άλλη προειδοποίηση δεν θα πάρετε για το ότι ε, τελειώνει ο χρόνο σα. Θα ήθελα επίση να υποδείξετε στην αρχή τη παρέμβασής σα ποιο υπουργό θα πρέπει να απαντήσει στην απάντησή σα, όχι τρει ερωτήσει σε ανά υπουργό μέσα στα πέντε λεπτά, γιατί δεν προλαβαίνετε να πάρετε την απάντηση. Παρακαλώ να είναι στοχευμένε οι ερωτήσει. Θα βοηθούσε αυτό. Ζητώ συγγνώμη που δεν ε, είμαι τόσο ευγενική και στρέφομαι και σε εσά, ε, Υπουργή. Θα είμαι αυστηρή και μαζί σα. Ε, έχετε κατανότατο όριο 7 λεπτά για τι εισαγωγικέ σα παρεμβάσει. Έχετε το χρονόμετρο εδώ δίπλα σα. Ζητώ συγγνώμη που ασχολούμαι με τέτοια πεζά πράγματα, αλλά αυτοί είναι οι κανόνε τη Επιτροπή. Αλλιώ δεν θα και αν έχετε κάποια παράπονα να κάνετε, να τα δείτε με τους αρμοδίους. Ο Υπουργός Σόιπλε θα αρχίσει. Παρακαλώ, Βόλφκα. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δίνετε να έχουμε μια ανταλλαγή απόψεων ε, να συζητήσουμε την Επιτροπή σας για την κατάσταση στη Γερμανία και περαιτέρω στην, στο Eurogroup και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Βέβαια, ο χρόνος είναι λίγος και θα ήθελα να σας ενημερώσω καταρχάς για την κατάσταση στη Γερμανία. Γνωρίζετε ότι και στη Γερμανία η οικονομία όπως και στην Ευρώπη και παγκοσμίως, έχει υποχωρήσει λίγο οικονομική δραστηριότητα. Την προπροηγούμενη εβδομάδα εγκρίναμε τον κρατικό προϋπολογισμό μας για το 2013. Ήδη από φέτος ανταποκρινόμαστε στις απαιτήσεις του Ευρωπαϊκού Παραγόγου Δικαίου ε, τηρούμε το όριο του ελλείμματος και σε όλα τα σημεία και στη διόρθωση ανισορροπιών ε, σύμφωνα με την έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προσαρμοστήκαμε και τηρούμε το κοινοτικό ευρωπαϊκό δίκαιο. Και σε ό,τι αφορά την κατάσταση στη Γερμανία θα ήθελα να περιοριστώ σε αυτή την περιγραφή. Στη Γερμανία έχει συζητηθεί κατά καιρού. Μήπως θα πρέπει τα ελλείμματα μας να τα μειώνουμε ε, με ταχύτερους ρυθμούς. Αλλά νομίζω ότι γενικότερα και στη μείωση του ελλείμματος, αλλά και στο δρόμο της εξισορρόπησης και της διόρθωσης των ανισορροπιών στην Ευρώπη, θα πρέπει να ακολουθούμε και τηρούμε το σωστό μέτρο και το σωστό ρυθμό. Στην, ε, στο Eurogroup την περασμένη εβδομάδα κάναμε σημαντικά βήματα και τώρα ε, συμφωνήσαμε και για την πληρωμή της επόμενης δόσης για το πρόγραμμα βοήθειας στην Ελλάδα. Ε, το επιτύχαμε. Στη Γερμανία η συζήτηση δεν ήταν εύκολη. Την περασμένη Παρασκευή συζητήσαμε την αλλαγή του μνημονίου για την Ελλάδα και δώσαμε την απαιτούμενη πρώτερη συμφωνία ε, της Γερμανικής Βουλής κατά πλειοψηφία με εξαίρεση μία πολιτική ομάδα στο Κοινοβούλιο. Όλες οι υπόλοιπες υπερψήφισαν ε, τις προϋποθέσεις για την εκταμείευση της επόμενης δόσης προς την Ελλάδα με όλες τις λεπτομέρειες στις οποίες δεν θα αναφερθώ ε, αυτή τη στιγμή περί τίνος πρόκειται σε αυτά τα θέματα. Αυτό που ενδιαφέρει εμάς και είναι ίσως ε, πιο σημαντικό να το πω γενικότερα, είμαστε πεπισμένοι ότι για να λύσουμε τα προβλήματα που έχουμε με το κοινό νόμισμα στην ΟΝΕ, στην Ευρώπη, αυτό πρέπει να γίνει βήμα-βήμα. Αλλά σε κάθε βήμα, και αυτό ισχύει και για τη συζήτηση που θα κάνουμε αύριο κυρίως στο ΕΚΟΦΗΝ, για την ενιαία τραπεζική εποπτεία. Σε κάθε βήμα θα πρέπει να προσέχουμε λοιπόν στην Ευρώπη ποιες είναι οι διαφορές ανάμεσα στα 17 κράτη που συμμετέχουν στην ΟΝΕ και στα 10 που ακόμα δεν συμμετέχουν στο κοινό νόμισμα. Λοιπόν, να μην διευρύνουμε το χάσμα κάθε φορά, αλλά να διατηρούμε το δρόμο ανοιχτό για ε, όλα τα υπόλοιπα δέκα ή όσα τα επιθυμούν για να μπουν στην ΟΝΕ. Να μην διευρύνονται λοιπόν τα χάσματα και ε, να μην χωρίζουν οι δρόμοι μας. Αυτό θα συζητηθεί και στο ΕΚΟΦΗΝ για την ενία τραπεζική εποπτεία και θα πρέπει να το έχουμε υπόψη μας. Σε ό,τι αφορά λοιπόν τη σταδιακή και βήμα-βήμα λύση ε, των προβλημάτων που έχουμε στην ΟΝΕ, είναι διπλή η προσέγγιση μας. Αφενός, μπορούμε να επιλέξουμε ένα δρόμο με προσαρμογές και μέτρα στα κράτη-μέλη και έχουμε κάνει σημαντικές πρόοδους. Την περασμένη Παρασκευή εξήγησα στη Γερμανική Βουλή και παρουσίασα όλα τα μέτρα που έχει λάβει η Ελλάδα και τις πρόοδους που έχει κάνει και στη βελτίωση των μακροοικονομικών της ε, δυνατοτήτων ανταγωνισμού ήδη τα όσα έχει επιτύχει. Θα πρέπει να συνεχιστεί αυτή η προσπάθεια. Αλλά δείχνει ότι ο δρόμος που έχει ε, ξεκινήσει δεν ειναι λανθασμενο λανθασμένος. Απλώς βήμα-βήμα θα πρέπει να προχωρούμε και να μην ε, δίνουμε λάθος κίνητρα σε λάθος ε, χρονική στιγμή. Θα πρέπει πάντα να έχουμε υπόψη μας τον ηθικό κίνδυνο, αλλά και να έχουμε συνέστηση του γεγονότος ότι χρειάζονται διαρθρωτικά μέτρα και είναι απαραίτητα αυτά για τον περιορισμό των ελλημάτων και αυτά γίνονται δεκτά μόνο εφόσον ε, διατηρείται η πίεση για δράση. Και αυτή η διαδικασία και η σταδιακή πρόοδος αφορά και την ε, επάνωδο της ε, εμπιστοσύνη των αγορών. Θεωρούν μίζωνα κίνδυνο την χρέωση των κρατών οι αγορές μετά την υπόθεση της Lehman Brothers και θεωρούν ότι η Ευρωζώνη έχει μεγαλύτερο κίνδυνο από άλλες περιοχές του κόσμου και οικονομίες που μπορεί να είναι πιο προβληματικές. Αυτό δείχνει λοιπόν πόσο περίπλοκη είναι η κατάσταση και στην ΟΝΕ και διεθνώς για την οικονομία, οι αγορές και οι φορείς της αγοράς και αυτοί πείθονται σταδιακά και βήμα-βήμα. Και αυτό πάλι λοιπόν δεν επιτυγχάνεται σε ένα και μοναδικό βήμα για να έχουμε μια καλύτερη δομή λήψης αποφάσεων μπορεί ε, να προχωρούμε ε, βάσει κειμένων συνθήκων και το κάναμε την τελευταία διετία με το Δημοσιονομικό Σύμφωνο, ε, το six το ΤΟΥΠΑΚ, το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο, όλα αυτά τα μέτρα. Αλλά ταυτόχρονα χρειαζόμαστε για, και για μεγαλύτερες θεσμικές αλλαγές τροποποίηση των συνθήκων. Η κυβέρνηση της Γερμανίας είναι πρόθυμη να το πράξει αυτό, αλλά ε, γνωρίζουμε ότι δεν μπορούμε να περιμένουμε τροποποίηση των συνθήκων που χρειάζονται και το χρόνο τους για να λύσουμε τα προβλήματα. Θα πρέπει και εκεί να δείχνουμε ρεαλισμό. Εμείς είμαστε πεπισμένοι και έρχομαι τώρα σε μια γενική παρατήρηση για να καταλήξω ότι μια βιώσιμη ανάπτυξη στην Ευρώπη και μια τέτοια πολιτική εν ώψη των παγκοσμίων ε, προκλήσεων θα την επιτύχουμε μόνο όταν έχουμε ε, ισχυρή δημοσιονομική ε, πολιτική. Γιατί έχουμε και τη δημογραφία μας, έχουμε και τις εξελίξεις στις αναδυόμενες χώρες και στις αναπτυσσόμενες χώρες. Για να παραμείνουμε στην κορυφή της κοινωνικής πυραμίδας στην ε, Ευρώπη και παγκοσμίω θα πρέπει να φέρουμε καινοτομία. Δεν θα πρέπει λοιπόν να χαλαρώσει η πίεση ε, και να πέσουμε σε αυτό τον πειρασμό δηλαδή ε, ε, για την επίλυση των διαρθρωτικών προβλημάτων και των ζητημάτων της καταπολέμησης του χρέους. Όπως προχωρήσαμε τελευταία διετία, οφείλουμε να προχωρήσουμε και στο μέλλον. Σας ευχαριστώ πολύ. Thank you Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Χωρίς να δαπανώ περισσότερο χρόνο, θα ακολουθήσει. Όχι ότι χαλάσαμε χρόνο τώρα με τη δική σας παρέμβαση. Ε, θα δώσω αμέσως το λόγο στον ε, Πιέρ Μοσκοβίτσι. Κυρίε και κύριοι βουλευτέ, κύριε Υπουργέ, κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ για αυτή την πρόσκληση που με χαρά αποδέχτηκα. Και εγώ χαίρομαι να έρχομαι σε αυτό το κοινοβούλιο που γνωρίζω καλά επειδή εκτελέσα το δύο θητείε και υπήρξα και για ένα διάστημα αντιπρόεδρο του για το αξιοσημείωτο έργο σας και για το ευρωπαϊκό έργο που επιτελεί το Ευρωκοινοβούλιο σε αυτές τις δύσκολες στιγμές. Δεν ξέχασα λοιπόν αυτή την εμπειρία με τις νέε αρμοδιότητες που ανέλαβα. Θα ήθελα και εγώ να μιλήσω πρώτα απ' όλα για την εθνική μας κατάσταση και μετά για το ευρωπαϊκό, την ευρωπαϊκή μας θεώρηση. Για τη Γαλλία λοιπόν για τι πιο πρόσφατε εξελίξει έχουμε μια οικονομική στρατηγική τρίπτυχη. Ε, επάλυψη του χρέου Ευρώπη και ανταγωνιστικότητα για να ε, διορθώσουμε τις βαθιές ανισορροπίες της γαλλική οικονομίας που έχει οξύνει η κρίση. Είναι σημαντικές τη ε, ισορροπία, διότι υπάρχει 10% ποσοστό ανεργία. Η ανάπτυξη είναι άτονη εδώ και πολλά τρίμηνα και το δημόσιο χρέος έχει φτάσει σε ένα επίπεδο το οποίο δεν μπορεί πλέον να αντιμετωπιστεί. Η διάγνωσή μας είναι ότι χρειαζόμαστε μια εύρωστη οικονομία με πλεονεκτήματα, με δυνατά σημεία, αλλά και ανταγωνιστικότητα εδώ και μια δεκαετία υποχωρεί. Αυτό λοιπόν μας οδηγεί στην τρίπτυχη λύση μας, την απάλληψη του χρέους πρώτα απ' όλα. Θα πρέπει η Γαλλία και πάλι να αναλάβει την τύχη στα χέρια της, την, την τύχη της χώρας. Δηλαδή θέλουμε να φτάσει το έλλειμμα στο 3% του ΑΕΠ μέχρι το 2015 13, να ξαναβρούμε τη διορθωτική ισορροπία μέχρι το 2017 και γι' αυτό σε έξι μήνες θα ε, προτείνουμε έξι δημοσιονομικά νομοσχέδια στο Γαλλικό Κοινοβούλιο προσπαθώντας να εξεύρουμε τη δημοσιονομική ισορροπία και προσπαθώντας να διατηρήσουμε την κοινωνική δικαιοσύνη. Δηλαδή να εξηγιανθεί η κοινωνική μας πολιτική. Έπειτα η Ευρώπη, δεύτερο σκέλος, με τους ε, Γερμανούς ε, εταίρους μας και χαίρομαι ιδιαίτερα που βρίσκομαι εδώ με τον κύριο Σόιμπλε για το λόγο αυτό. Προσπαθούμε να καταρτήσουμε μια ευρωπαϊκή στρατηγική με τέσσερι προτεραιότητε. Πρώτα απ' όλα, επίλυση τη κατάσταση των χωρών με δυσχέρειε. Η συμφωνία που επεγράφει για την Ελλάδα την περασμένη εβδομάδα με πολλή δυσκολία, αλλά με αποφασιστικό τρόπο είναι μια, ένα σημείο καμπή και για την Ελλάδα και για την Ευρωζώνη επίσης, διότι να θα επιτρέψει να δημιουργηθούν όροι εμπιστοσύνη και ίσως και ανάπτυξης. Δεν επιλύονται βέβαια έτσι όλα τα προβλήματα, αλλά θα επηρεαστεί η εθνική κατάσταση. Έπειτα η Τραπεζική Ένωση. Επειδή ακριβώς ε, υπάρχει αυτή, αυτός ο συσχετισμός μεταξύ δημόσιο χρέους και ε, τραπεζικού, προσπαθούμε ήδη να εξεύρουμε λύσεις με νομοθετικές προτάσεις που θα έχουν ήδη ολοκληρωθεί στο 2012. Ε, για, το, για την Ευρώπη επίσης και την ανάπτυξη θα πρέπει να υπάρξει και ένα σχετικό σύμφωνο ανάπτυξης με ένα πρόγραμμα για την Ευρωζώνη πιο συγκεκριμένο. Δεύτερος πυλώνας της στρατηγικής μας είναι η ανταγωνιστικότητα. Ο πρωθυπουργό μα και ο πρόεδρο τη ε, Δημοκρατία, τη Γαλλική Δημοκρατία, ε, δήλωσαν ότι θα δημιουργηθεί ένα σύμφωνο ανταγωνιστικότητα που αύριο θα ανακοινωθεί επισήμω στην ε, Γαλλία, ώστε οι επιχειρήσει να διαθέτουν ένα περιθώριο λιγμών για να επενδύουν και να κάνουν προσλήψει. Με σκοπό να μεταρρυθμιστεί και η αγορά εργασία, κάτι που θα έχει ιστορική σημασία στην Γαλλία και να μπορέσουμε να φτάσουμε στο σημείο να πούμε ότι η Γαλλία μπορεί να κατακτήσει και πάλι ε, ένα σημαντικό μερίδιο στην αγορά και μια σημαντική θέση ως προς την ανταγωνιστικότητα. Τώρα για την Ευρωζώνη. Για το πώς συμπεριλαμβάνουμε τη διάσταση Ευρώπης στην εθνική μας στρατηγική. Η Ευρωζώνη είναι ένα οικοδόμημα θαυμάσιο. Αλλά ημιτελέ η κρίση έχει δείξει ακριβώς τι μας έλειπε. Μηχανή, μηχανισμοί σταθερότητας σε περίπτωση ασυμμετρικών προβλημάτων ή ετερογένεια στη διαχείριση των προβλημάτων και δυσκολία να ληφθούν γρήγορες αποφάσεις και εύληπτες. Ε, εδώ πέρα το νήμα που συνδέει όλα αυτά τα στοιχεία είναι η αλληλεγγύη. Η ευρωπαϊκή κρίση είναι μια κρίση ολοκλήρωσης. Ε, είναι έλλειμμα Ευρώπης και δυσκολια να ληφθουν γρηγορες αποφασεις και ε εδω περα το νημα που συνδεει ολα αυτα τα στοιχεια πλεόνασμα το πρόβλημα. Εδώ λοιπόν θέλουμε να συμπληρώσουμε την Ευρωζώνη, να την προοικοδοτήσουμε με τα μέσα ώστε να αντιμετωπίσει τα προβλήματα και αυτό βάσει της αλληλεγγύης. Θα γίνουν κάποιες συγκεκριμένες προτάσεις με, δημοσιονομική με ίδιους πόρους, ε, με διαφορετική από τον προπολογισμό των 27, αντιμετώπιση των αντικυκλικών φαινομένων, και χρηματοδότηση δράσεων για σημαντικά ζητήματα όπως η κοινωνική δράση, η ανταγωνιστικότητα ή ένα κατόφλι για την αντιμετώπιση τη ανεργία στην Ευρωζώνη. Έπειτα, τα ομόλογα χρέου στην Ευρωζώνη από κοινού και βεβαίως η ε, δημοκρατική νομιμοποίηση των αποφάσεων που λαμβάνονται στο επίπεδο τη Ευρωζώνη. Διότι μέχρι τώρα το μοντέλο μα δεν λειτουργεί. Υπάρχει διάσταση των Εθνικών Κοινοβουλίων και από την άλλη ε, του Ευρωκοινοβουλίου. Γιατί να μην υπάρξει μια επιτροπή που να εκλέγεται από τους πολίτες της Ευρωζώνης με νομοθετικό ρόλο, εφόσον δεν υπάρχει υπολογισμό της Ευρωζώνης. Επίσης, μεσοπρόθεσμα, Νομίζω θα πρέπει να υπάρχει και εκτελεστική εξουσία στην ε, Ευρωζώνη, στο πρόσωπο ενός Υπουργού, ο οποίος θα μπορεί εμέσως ή αμέσως να ανελάβει αρμοδιότητες ε, ξενόματος των Ευρωπαίων πολιτών της Ευρωζώνης. Αυτός ο μηχανισμός αλληλεγγύης και εφόσον θεσπιστεί στην Ευρωζώνη θα πρέπει να λειτουργεί και εύρυθμα, με αυστηρότερα μέτρα, στο δημοσιονομικό επίπεδο, ώστε λόγου χάρη η κοινή έκδοση χρέου να ελέγχεται και ενδεχομένω να γίνει και αναθεώρηση των συνθήκων εφόσον χρειαστεί. Δεν είμαι αντίθετο με αυτή την ιδέα, αλλά θα πρέπει να φανεί πώ θα γίνει αυτό. Πρώτα απ' όλα λοιπόν θα πρέπει να έχουμε εξηγέννηση, μετά την διακυβέρνηση και μετά να δούμε μακροπρόθεσμα τι θέλουμε. Έτσι θα μπορέσουμε να ανακτήσουμε την εμπιστοσύνη των πολιτών μα ενδεχομένω και αυτέ είναι κάποιε πρώτε ιδέε. Έχουμε μια προθεσμία για να συζητήσουμε αυτές τις βασικές ε, ιδέες. Το Δεκέμβριο το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο που θα συζητήσει αυτές τις πρώτες αυτά τα πρώτα σχέδια και έως το 2014 μας μένει περίπου ένας χρόνος για να αποσαφινιστεί το πολιτικό αυτό σχέδιο που θέλουμε να το γνωστοποιήσουμε και στους πολίτες και να έχουμε αρκετή νομιμοποίηση δημοκρατική ώστε να μπορέσουμε να ενισχύσουμε τις αποφάσεις αυτές που θέλουμε να φέρουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και η Γαλλία ακριβώς θα συνεργαστεί, ε, θα εργαστεί μάλλον σκληρά για την δημοκρατική αυτή ολοκλήρωση, όπως ε, έχει δείξει ο Γάλλος Πρόεδρος και η κυβέρνησή του. Σας ευχαριστώ. Θα περάσουμε ευθύ αμέσω σε ερωταπαντήσει. Πρώτη ερώτηση από πλευράς του ΕΛΚΑ. Παμπλό Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να ρωτήσω τον Υπουργό, κύριε ε, Σόιμπλε. Εγώ ζω στη Βόρεια Ισπανία Εκεί οι επιχειρήσεις δεν μπορούν να χρηματοδοτηθούν από τη μια πλευρά των σύνορων στην Ισπανία έχουν πολύ ε, δύσκολη δανειοδότηση. Από την άλλη πλευρά των σύνορων ε, στη Γαλλία είναι σχεδόν ε, δωρεά η χρηματοδότηση. Αυτό είναι ένα πρόβλημα ανταγωνιστικότητα. Αυτό θα λυθεί μόνο όταν επέλθει η Τραπεζική Ένωση. Πιστεύετε κύριε Υπουργέ ότι η Κυπριακή Προεδρία αύριο θα λάβει την εντολή για να αρχίσει διαπραγματεύσει με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που ήδη έχει γνωμοδοτήσει και ξεκάθαρα ε, στις εκθέσεις ε, Tyson και Giggold έχει λάβει θέση. Και αν η Κυπριακή Προεδρία λάβει αυτή την εντολή, ποια θα είναι τα βασικά στοιχεία της συμφωνίας. Ευχαριστώ κύριε Υπουργέ. Wolfgang, νομίζω ότι απευθυνόταν το ερώτημα σε σένα. Ευχαριστώ πολύ. Νομίζω ότι στην τραπεζική εποπτεία έχουμε δύο ζητήματα που ελπίζω να λυθούν, αλλά δεν είμαι βέβαιος ότι αύριο θα καταλήξει το ΕΚΟΦΕΝ σε εντολή. Το πρώτο είναι το θέμα της διακυβέρνησης και πιστεύουμε ότι ε, αυτό που έχει αποφασιστική σημασία είναι Δύο σημεία, τα οποία ανέφερα προηγουμένως. Θα πρέπει ε, ε, να υπάρχει σαφής διαχωρισμός ανάμεσα στην νομισματική πολιτική και στην τραπεζική εποπτεία για να διαφυλαχθεί η ανεξαρτησία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Και επίσης θα πρέπει να βρούμε μια ρύθμιση έτσι ώστε ε, και τα μη μέλη της Ευρωζώνης να έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν. Το είπαν αυτό οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων. Επίσης όρις να συμμετέχουν στην τραπεζική εποπτεία και μη μέλη της Ευρωζώνης. Δεν ξέρω εάν θα βρούμε αύριο λύση. Δεν μπορώ να το προεξοφλήσω. Επιτρέψτε μου όμως να κάνω ένα δεύτερο σχόλιο. Έχω την εξή εντύπωση οι προσδοκίες ε, από τη τραπεζική εποπτεία για τη χρηματοδότηση των επιχειρήσεων νομίζω είναι λίγο υπερβολικές. Ε, θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι η απόφαση της 29ης Ιουνίου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου ήταν αυτή τη στιγμή ε, λειτουργεί η τραπεζική εποπτεία με συγκεκριμένες προϋποθέσεις να υπάρχει ένας διαχωρισμός ανάμεσα στον κίνδυνο που αναλαμβάνουν οι τράπεζες ε, για τη χρηματοδότηση του κρατικού χρέους με ανακεφαλαιοποίηση ε, να υπάρχει δυνατότητα ε, ανάληψης από το μηχανισμό σταθερότητας. Δηλαδή να ζητάει ένα κράτος ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών, αλλά μαζί με το κράτος αυτό να συμφωνείτε ένα πρόγραμμα προσαρμογών. Αυτό δεν καταργείται. Αν θέλαμε να το καταργήσουμε, θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι θα ε, ε, εξαντλεί το πάρα πολύ γρήγορα ο μηχανισμός σταθερότητας, ο ESM εάν ε, απλούστατα ανακεφαλαιοποιούσαμε τις τράπεζες χωρίς προϋποθέσεις. Δηλαδή το, θα έλειωνε αυτό, θα εξαφανιζόταν. 80 δισεκατομμύρια ήταν το κεφάλαιο. Δηλαδή τόσο γρήγορα δεν λιώνουν τα χιόνια την Άνοιξη ούτε στα Πυρηναία ούτε στις Άλπεις. Θα είχε εξαντληθεί το ποσό αυτό ήδη από το 2014. Είδαμε από την τραπεζική κρίση τι έγινε το 2008. Στη Γερμανία και μόνο έχουμε συγκρίσιμα μεγέθη. Το 2008 χρειάστηκε να κεφαλοποιήσουμε τις τράπεζές μας και θα πρέπει να βρούμε βρούμε στο μηχανισμό σταθερότητας, στο ESM, ότι αυτό είναι ένα τείχος προστασίας ε, ε, αλλά δεν, δεν προστατεύει υπερβολικά από νέα προβλήματα της χώρας. Παρακαλώ, προειδοποιώ να μην είναι υπερβολικές εκεί οι προσδοκίες μας. Ε, ο Παύλο, νομίζω έχω ένα λεπτό συμπληρωματικό. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή επιτευχθεί συμφωνία και μακάρι να ανατεθεί αυτή η εντολή στην Κυπριακή Προεδρία. Θα υπάρχει δυνατότητα άμεσης ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών. Ευχαριστώ, Υπουργέ. Ε, Μα σα είπα και προηγουμένω, όχι, δεν είναι άμεσο αυτό, δεν είναι αυτόματο. Θα πρέπει καταρχά, αυτή τη στιγμή δοθεί η εντολή και ολοκληρωθεί ε, το νομοθετικό πλαίσιο θα χρειαστεί κάποιο χρόνος. Και επίσης το 2013 θα στηθεί αυτή η τραπεζική εποπτεία. Λοιπόν, και για να λειτουργήσει, για να αρχίσει να λειτουργεί θα χρειαστεί χρόνος. Από εκεί και πέρα θα υπάρχει δυνατότητα άμεσης ανακεφαλοποίησης, αλλά πάντα με τις ισχύουσες συνθήκες και προϋποθέσεις για να καταβληθεί ένα ποσό από το ESM. Αυτό παραγνωρίζεται κατά καιρού και παρακαλώ να μην το παραγνωρίζουμε γιατί δημιουργούμε φρούδες ελπίδες. Η Ισπανία δεν μπορεί να περιμένει τόσο καιρό. Υποθέτω ότι στην Ευρωζώνη θα μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε αυτή την απόφαση και ε, για την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών από χρήματα του ESM μέσω όμως του Ισπανικού κράτους Γι' αυτό καλό να μην συνδέουμε υπερβολικέ προσδοκίε, ότι με μια τέτοια εντολή θα είχαν άμεση πρόσβαση οι τράπεζε. Δεν είναι μόνο προθύστερο αυτό, είναι και υπερβολικό ω παραδοχή. Σας ευχαριστώ. Θα αφήσουμε το χρονόμετρο την επόμενη φορά για να γνωρίζουμε και αν ε, τηρείται ο χρόνος ομιλίας. Η Ελίζα τώρα. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να απευθύνω και εγώ το ερώτημά μου προς τον Υπουργό Σόιμπλε. Θα θέλαμε να σε ευχαριστήσουμε για τη σημερινή σας παρουσία. Τρία σύντομα ερωτήματα έχω. Πρώτον, η Γερμανία τηρεί απαρέγκλητα τη νομική βάση για όλες τις δημοσιονομικές παρεμβάσεις, θα ήθελα να ρωτήσω. Υπάρχει πρόβλημα με την νομική βάση της Τρόικα, δηλαδή παρεμβαίνουν αυτή τη στιγμή στις χώρες μας, σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Δεύτερον, ε, προ προς τις συνταγές που ακολουθούμε, ποιο είναι το αποτέλεσμα. Κάνουμε πλημελείς υπολογισμούς, γιατί χρησιμοποιούμε πλημελείς συντελεστές και Και λένε κάποιοι αυτή τη στιγμή ότι με την ε, υπάρχουσα νομική βάση, αν χρησιμοποιήσουμε όλο το διαθέσιμο περιθώριο του six-pack και, της και του Δημοσιονομικού Συμφώνου, θα μπορούσαμε να αναμένουμε καλύτερα αποτελέσματα παρατείνοντας ε, το χρόνο της άσκησης ε, της δημοσιονομικής πειθαρχίας. Συμφωνείτε ή όχι με αυτό. Ευχαριστώ. Wolfgang, για σένα και πάλι Πιστεύω ότι η Τρόικα τηρεί αυστηρά την εντολή της κατά τη διάρκεια των εργασιών της. Δεν έχω ποτέ διαπιστώσει κάτι που να μας κάνει να αμφιβάλλουμε. Εμείς παρακαλέσαμε την Τρόικα να παρέμβει στο μηχανισμό διάσωσης. Πρώτα το EFSF και μετά το ESM. Είναι τρεις ανεξάρτητες δομές και θεσμικά όργανα, κάνουν εκθέσεις και διαπραγματεύσεις βεβαίως με το εκάστοτε κράτος μέλος και πιστεύω ότι η Τρόικα ανταποκρίνεται ε, θαυμάσια στις προϋποθέσεις αυτές και στην εντολή της. Στη συνέχεια, νομίζω ότι η πολιτική αυτή είναι επιτυχής. Έχουν σημειωθεί σημαντικές στην Ιρλανδία και την Πορτογαλία που είναι σε πρόγραμμα. Η Ιρλανδία έχει πάρει το δρόμο προς τις αγορές και η Πορτογαλία είναι σε καλό δρόμο. Τα προγράμματα είναι τακτά και σωστά. Έχουμε ένα ειδικό πρόβλημα στην Ελλάδα που μας έχει απασχολήσει εντατικά, αλλά όπως είπα προηγουμένως, την περασμένη Παρασκευή εξήγησα στη Γερμανική Βουλή στην Bundestag και παρουσίασα όλα τα επιτεύγματα της Ελλάδας. Και βέβαια, επίσης, είπα ότι στο μεταξύ όλοι μαζί καταλάβαμε, ίσως περισσότερο από ό,τι πριν από τρία χρόνια, πόσο βαθιά είναι τα προβλήματα της Ελλάδας, που στη δημόσια συζήτηση σε πολύ μεγάλο βαθμό έχουν υποτιμηθεί. Και πολύ περισσότερο ακόμα και στην Ελλάδα, την ίδια, για το τι πρέπει να κάνει η Ελλάδα. Σύμφωνα με την άποψη πολλών οικονομολόγων, και σε μια νομισματική ένωση αυτό συνδέεται με τεράστιες ε, προσπάθειες και στην εσωτερική πολιτική και τεράστιες πιέσεις. Εξού και η συζήτηση τις τελευταίες εβδομάδες με την Τρόικα και ιδιαίτερα με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Ε, είχαμε εντατικότατες ε, διαβουλεύσεις. Αλλά επαναλαμβάνω ότι πιστεύω ότι και η Ελλάδα είναι στον ορθοδρόμο. Εάν καταφέρει να συνεχίσει με συνέπεια αυτό το δρόμο τελικά θα επιτύχει. Και στα άλλα κράτη-μέλη αυτό συμβαίνει. Στην Ισπανία έτσι κι η κατάσταση είναι ιδιάζουσα. Έχει ιδιαίτερα προβλήματα ε, στον τραπεζικό τομέα και με εξαίρεση αυτά που έχουμε βρει κάποια λύση περισσότερα είναι αυτά τα προβλήματα τα τραπεζικά παρά τα ε, ειδικά πραγματικά προβλήματα της οικονομίας με κίνδυνο μετάδοση σε άλλες χώρες. Δεν σας ακούει. Ένα λεπτάκι σταματήσαμε το χρονόμετρο, Υπουργέ. Καταλαβαίνω αυτά που λέτε. Όμως η ανεργία σε κάποιες χώρες ε, έχει φτάσει το 50% των νέων ε, και σε πολλούς ε, δημιουργείται ένας πολύ άσχημος φαύλος κύκλος και ταυτόχρονα οι καλύτερες οικονομίες που εκπροσωπούνται εδώ δεν θα γνωρίσουν αύξηση άνω του 1%. Ποιο είναι το μέλλον της Ευρώπης. Κάτι πρέπει να αλλάξει. Ευχαριστώ. Είναι γεγονός. Αλλά το θέμα είναι ποια είναι η αιτία και ποιο είναι το αποτέλεσμα. Μπορεί να διαφωνούμε στο θέμα του αιτίου και του αιτιατού, του αιτίου και της συνέπειας. Εμείς ε, θεωρούμε ότι η βιώσιμη ανάπτυξη μπορεί να επιτευχθεί μόνο με το δρόμο που σας παρουσίασα εισαγωγικά. Και κατά τα άλλα πιστεύω ότι εάν εφαρμοστεί και στην Ισπανία και σε άλλες χώρες θα οδηγήσει σε επιτυχία. Επίσης γνωρίζω ότι η μεγάλη ανεργία των νέων σε πολλές χώρες είναι μεγάλο πρόβλημα και με την Ισπανία είμαστε σε ε, στενή ανταλλαγή απόψεων για να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε ευρωπαϊκά βράχη πρόθεσμα σε διμερές επίπεδο για να βοηθήσουμε και σε αυτή την κατεύθυνση. ευχαριστώ. Βολφ Ευχαριστώ. Καταρχάς μια ερώτηση προς εσάς κύριε Σόιμπλε, κύριε Υπουργέ η Ευρώπη αντιλαμβάνεται τον εαυτό της ως ε, ένωση αξιών και αξία σημαίνει ότι και τα κράτη και τα πρόσωπα πρέπει να φέρονται αξιοπρεπώς ο ένας τον άλλον ε, διότι έχουμε πραγματικά αμαρτάνει ε, ε, ε, μια μεγάλη γερμανική λαϊκή εφημερίδα όταν μιλάει για τους Έλληνες του λέει οι Έλληνες της χρεοκοπίας και με ενοχλεί επίσης στην Ελλάδα στις διαδηλώσεις όταν εμφανίζουν την καγκελάριο ως SS, με στολή SS. Πώς είναι αυτή η επικοινωνία μεταξύ πολιτικών και πολιτών. Πώς ε, βλέπετε τις δυνατότητες βελτίωσης και αλλαγής αυτών των καταστάσεων. Και στα γαλλικά τώρα μια ερώτηση για εσάς κύριε Υπουργέ Μοσκοβισή. Τις εξής δύο. Για το πρόγραμμα ε, αγοράς του, εξαγοράς του κρατικού χρέους στην χώρα που έχουμε πρόβλημα στην Ευρωζώνη. Για την, ε, για την πολιτική λοιπόν ένωση. Είναι φανερό εξ αρχής ότι το ευρώ δεν μπορεί να πετύχει εάν δεν υπάρξει πραγματική πολιτική ένωση στην Ευρωζώνη. Το θίξατε νομίζω, αλλά κάποιοι πρώτα ζητούν την αλληλεγγύη και μετά τη μετατροπή της Ευρωζώνης σε μια μορφή πολιτικής ένωσης. Ενώ άλλοι λένε ότι χρειάζεται το αντίστροφο. Πρώτα πολιτική ένωση και μετά αλληλεγγύη. Εσείς τι γνώμη έχετε. Πρέπει να μοιράσω το χρόνο. Βόλφανγκ, θα πάρεις πρώτος το λόγο, αλλά δυόμιση λεπτά σε παρακαλώ για να προλάβουμε για δεύτερο ερώτημα. Θα αφήσω το περισσότερο χρόνο στον Πιέρ. Κύριε Κλίντς, ανέκαθεν, ήδη πριν από δυόμιση χρόνια έλεγα στη Γερμανική Βουλή ότι θα πρέπει να σεβόμαστε τις θυσίες του ελληνικού λαού. Ξέρουμε ότι οι είναι ταραγμένοι και ε, αναγκαίες είναι και οι διαδηλώσεις και ένα τμήμα του τύπου υπερβάλλει και όλοι υφίστανται τις συνέπειες. Και εγώ είχα την τιμή να εμφανιστώ με στολίες στις ελληνικές εφημερίδες. Αλλά ταυτόχρονα συναντώ πολλούς Έλληνες στον δρόμο που μου ευχαριστούν για τις προσπάθειες που καταβάλουμε. Δεν θα σταματήσει η γερμανική κυβέρνηση υπεύθυνα να εξηγεί τι είναι εφικτό και για ποιο λόγο και επίσης να επισημαίνει ότι στην Ελλάδα για τον κόσμο, για τους ανθρώπους είναι τεράστια η πίεση. αυτό που έχει αποτύχει στην Ελλάδα είναι η ελίτ, αλλά δεν μπορούμε να το αλλάξουμε. Oui, sur, sur για την επαναγορά κρατικού χρέους, το debt buyback, όπως λέγεται, δεν ανησυχώ ιδιαίτερα. Ξέρουμε ποια είναι η πρόθεση των ελληνικών αρχών από τη μια τι είδου συμβουλέ του παρέχονται. Μιλάμε για οργανισμού που θα πουλήσουν το χρέο το οποίο διαθέτουν, ε, έχουν στην κατοχή του στο 30% τη αρχική του αξία. Νομίζω ότι με την Ελλάδα θα την κερδίσουμε αυτή την πρόκληση μαζί. Ε, την Παρασκευή η κυρία Λαγκάρ ήταν στο Παρίσι και συζητήσαμε. Ήταν αρκετά αισιόδοξη για το πώ θα λειτουργήσει ο μηχανισμό. Απλώ πρέπει όλα να γίνουν γρογά, γιατί θα πρέπει η απόφαση στι 13 Δεκεμβρίου να εκτελεστεί άμεσα για άμεση εκταμείευση. Θα πρέπει να είμαστε κυριαλιστές και ελπίζω όλα να λειτουργήσουν σωστά. Για την πολιτική ένωση τώρα κατά τα άλλα, αυτό που είπε και ο πρόεδρο τη Γαλλική Δημοκρατία είναι ότι χρειαζόμαστε ολοκλήρωση δημοκρατική. Και στη δημοσιονομικό επίπεδο και στο κοινωνικό Διότι αλληλεγγύη θα πρέπει να φτάσει στα όρια της. Δηλαδή, με την συνταγματική συνθήκη βρισκόμουν σε αυτή την ε, αίθουσα ως ε, βουλευτής και Είδαμε τι έγινε με το δημοψήφισμα στη Γαλλία. Βλέπουμε ότι ως προς την αλληλεγγύη λοιπόν η Ευρώπη δεν προχωρά με, με ίσο ρυθμό. Κάποιοι θέλουν από τη μια την σταθεροποίηση και άλλοι την αλληλεγγύη. Θα πρέπει λοιπόν αυτά τα δύο σκέλη να φροντίσουμε να προχωρούν και να συμβαδίζουν. Σας είπαμε ότι στη γαλλική πολιτική το πρώτο στοιχείο είναι η απέλευση του χρέους. δεν είναι χαλαρή στην πολιτική της η Γαλλία με μελλοντολογικές ε, θεωρήσεις. Θα πρέπει να προχωρήσουμε με τα δύο αυτά σκέλη, σταθεροποίηση και αλληλεγγύη, μαζί με τη Γερμανία. Ευχαριστούμε. Αυτή ήταν η προειδοποίηση για τα 30 δευτερόλεπτα. Καλά τα καταφέρατε από τους συντηρητικούς ε, και η Swimmer. Παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να απευθύνω στο Γάλλο Υπουργό, αν μου επιτρέπετε τις ερωτήσεις μου. Ε, στο Τόκιο σήμερα το πρωί ο Κρίσταν Νόιερ, που είναι επικεφαλής της Banque de France, Μεταξύ άλλων είπε ότι οι κυβερνήσεις της Ευρωζώνης πρέπει να αναβαθμίσουν τα δημοσιοοικονομικά και να προβούν σε διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις ώστε να καταστούν οι περιφερειακές αυτές οικονομίες ε, πιο ανταγωνιστικές. Άρα υπονοεί ότι μπορούν να γίνουν περισσότερα πράγματα. Στα εισαγωγικά στα σχόλια μας μιλήσατε για μείωση του διαρθρωτικού ελλείμματος. Όμως ε, στους επενδυτές ε, υπάρχουν πολλοί αποκλίνουσες απόψεις ανάλογα με το αν σκέφτονται χωρίς ή με προβλήματα. Πιστεύετε στη μακροπρόθεσμη ανταγωνιστικότητα. Πιστεύετε ότι μακροπρόθεσμα συγγνώμη, η Ευρώπη θα προσελκύσει επενδύσει. Χάρη στην ερώτησή σας μπορώ να σχολιάσω διεξοδικότερα την κατάσταση στη Γαλλία. Είπα ήδη ότι είναι κρατεά η οικονομία σταθερή με ισχυρά του που γνωρίζετε όλοι. Είναι μεγάλη η οικονομία, διαφοροποιημένη, ποιοτικές υπηρεσίες, ε, υποδομές, ε, υψηλή ειδίκευση. Αλλά ταυτόχρονα τα τελευταία δέκα χρόνια έχει απολέσει μεγάλο κομμάτι της ανταγωνιστικότητας, 10% ανεργία. 91% του ΑΕΠ το δημόσιο έλλειμμα, το εμπορικό έλλειμμα, έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου 170 ε, ε, ε, δισεκατομμύρια σε εμά έναντι 160 πλεονάσματος στην Γερμανία. Πρόβλημα στη βιομηχανική παραγωγή. Αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι από κοινού να αντεπεξέλθουμε σε αυτές τις δυσκολίες ε, με τρόπο ώστε να ανακάμψουν τα δημοσιοοικονομικά, μείωση του χρέους και του ελλείμματος όπως σας έλεγα προηγουμένως, βελτίωση της παραγωγικής μας μηχανής ε, και ανάκαμψη επίσης στον κοινωνικό τομέα και πανέρχομαι τώρα στο τρίπτυχο, την γαλλική πολιτική, δηλαδή εμπιστοσύνη στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην Ευρωζώνη και τέλος ανταγωνιστικότητα. Ε, οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις που ζητούν κάποιοι από τη Γαλλία. Τώρα αποφασίσαμε να τις δρομολογήσουμε διότι πέρα από τα φορολογικά κίνητρα στα οποία αναφέρθηκα έχουμε ένα φορολογικό πρόγραμμα 35 μέτρων για ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, ε, σταθερότητα, εξυγχρονισμός της διοίκησης, ε, πλούστευση των σχέσεων με τις μικρο, ε, μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ενθάρρυνση της έρευνας, βελτίωση της κατάρτισης και ούτω καθεξής. Αποφασίσαμε να αντιμετωπίσουμε κατάματα όλες αυτές τις δυσκολίες και να προβούμε και στην μεταρρύθμιση αγοράς-εργασίας. Ε, τώρα γίνεται διαβούλευση με τους κοινωνικούς εταίρους ε, για να ε, καταστήσουμε ασφαλέστερες τις θέσεις απασχόλησης και ταυτόχρονα θα μειώσουμε τον επισφαλή χαρακτήρα των θέσεων εργασία. Αυτό περνάει μέσα από την εκάστοτε σύμβαση εργασία, αλλά ταυτόχρονα να ενισχύσουμε την παραγωγική μα μηχανή προσδίδοντα μεγαλύτερη ευελιξία για να χειριστούμε τι μελλοντικέ δυσκολίε μα. Είναι συνεκτικό το πλαίσιο που προτείνουμε, Α αποφύγουμε όμω στα στερεότυπα. Είναι ελκυστική ήδη η Γαλλία για, τη, για τους Νομίζω είμαστε στη δεύτερη θέση στην Ευρώπη. Δεν νομίζω ότι ε, θα πρέπει να μας λυπάται κανείς. Δεύτερον, για τη χρηματοδότηση του χρέου μας ε, είναι πολύ χαμηλά τα επιτόκια που μας ζητάνε και αυτό σχετίζεται με την ποιότητα του δημοσίου χρέους και τον τρόπο με τον οποίο το διαχειριζόμαστε. Αλλά είμαστε πιο επιθετικοί στην πολιτική μας. Ε, δηλαδή, στην επόμενη πενταετία με την καταπολέμηση της ανεργία ε, και ε, την αποκλιμάκωση του χρέου, τη βελτίωση των δημοσιοοικονομικών ε, και τη μείωση του τμήματο του ελλείμματο στο δημόσιο ΕΕΠ θα τονώσουμε την ανταγωνιστικότητα και θα ενισχύσουμε την βιομηχανική παραγωγή τη Γαλλία. Χρειάζεται χρόνο, βέβαια και το 2013 θα είναι δύσκολο έτος γιατί ταυτόχρονα πρέπει να κάνουμε μια προσπάθεια 30 δισεκατομμυρίων για τη μείωση του ελλείμματο ενώ είναι παραπέει λίγο η ανάπτυξη ανάπτυξη, αλλά αυτήν τη στρατηγική προκρίνουμε και θα την οδηγήσουμε ε, μέχρι το τέλος. Σάρων Πόλης και σε παρακαλώ γρήγορα. Είναι μία επερώτηση, ε, θα ξέρουν όλοι ε, την απάντηση, αλλά εν πάση περιπτώσει νομίζετε ότι οι οργανισμοί εξολόγηση πιστοληπτικής ικανότητας κάνουν λάθος απάντηση. Ε, υπάρχει μία που κάνει μάλλον θετικές ε, αποτιμήσεις, ε, η άλλη διατήρησε μάλλον υψηλά την ε, βαθμολογία. Τι να κάνουμε, αυτές έχουμε. Ε, από πλευράς των Πρασίνων, Ζαν Πολβεζέ. Ε, ερώτησή μου απευθύνεται στον Γάλλο Υπουργό Οικονομικών. Κύριε Μοσκοβισή, θα μπορούσατε να μας διαφωτίσετε για την τραπεζική μεταρρύθμιση που η γαλλική κυβέρνηση θέλει να υλοποιήσει γοργά κιόλα. Νομίζω το νομοσχέδιο θα εξεταστεί από το Συμβούλιο των Υπουργών πριν το τέλος της χρονιάς. Κάτι που αντιφάσκε με την όλη σκέψη της, ε, που υπάρχει στην Ευρώπη για την Τραπεζική Ένωση. Και επίση συσχετίζοντα το θέμα με το εξή, ε, συσχετιζόμενο με το εξή, μιλάτε για μια σημαντική μεταρρύθμιση που σκοπό θα έχει την εξυγίανση του τραπεζικού τομέα. Αυτό φαίνεται να ισχύει με το νέο καθεστώς ευρωπαϊκής λύσης σε περίπτωση κρίση. τη λύση εκαθάρισης ε, των τραπεζών και την προληπτική εποπτεία. Πώς θα γίνει ο διαχωρισμό όμως της καταθέσεις ε, και της αναλήψης τράπεζες από τη μια ε, και το τι συμβαίνει με τις ε, δράσεις του στην αγορά, στις αγορές Και επίσης για την έκθεση Λικάνεν. Οι λεγόμενες δράσεις και οι θέσει στην διατραπεζική αγορά πώς θα διαρθρωθούν με την τραπεζική αυτή μεταρρύθμιση. Μήπως διατηρείται το status quo και ουσιαστικά διατηρείται η σύγχυση και διονύζεται ο κίνδυνος. Καλά ξεκινήσατε την ερώτηση. Είναι λιγότερο θετικό το τέλος της. Να σας πω κύριε Μπεσέ ότι όχι. Θέλουμε να αναλάβουμε ακριβώς την δέσμευση του Γάλλου πρόεδρο της Δημοκρατίας κατά την προεκλογική του εκστρατεία με τον διαχωρισμό και την αντιμετώπιση της κερδοσκοπίας. Ο κίνδυνος που αναλαμβάνουν οι τράπεζες, στις ε, δράσεις του στην αγορά, θα πρέπει να είναι ανάλογος με τις ανάγκες χρηματοδότησης της οικονομίας. Γι' αυτό θα παραμένουμε κοντά στις συστάσεις της έκθεσης Λικάνεν, ε, με τον οποίο συζήτησα αυτοπροσώπως πριν από λίγες εβδομάδες, με στόχο οι δράσει στι αγορές να μην επηρεάσουν τι σχέσεις με τους πελάτες και την εξυπηρέτηση του κοινού. Γι' αυτό οι θηγατρικέ trading ούτω ή άλλω έχουν μια πολύ ευρία περίμετρο στην έκθεση Λικάνεν. Γι' αυτό θα πρέπει να γίνει ο διαχωρισμό με τις δράσεις ακριβώς στις χρηματοπιστωτικέ αγορές. Εμεί θέλουμε κάτι πιο πραγματιστικό να μας επιτρέψει να διαχωρίσουμε την κερδοσκοπία από την πραγματική οικονομία. Θα είναι αρκετά ριζοσπαστική μεταρρύθμιση με την ενίσχυση τη εποπτεία, τη δυνατότητα λήψη αποφάσεων, την, τον διακανονισμό, το trading υψηλή συχνότητα, τι συναλλαγέ τη αγορά πρώτων υλών. Ίσως χρειαζόμαστε στη Γαλλία μια ιδιαίτερη τραπεζική δομή, εφόσον έχουμε και 4.000, 4 εκατομμύρια θέσει εργασία, 400.000 ε, θέσει εργασία στον τραπεζικό τομέα, θέλουμε λοιπόν το μοντέλο αυτό να αλλάξει. Θέλουμε να επιβιώσει της οικονομικής κρίσης με καλύτερο τρόπο κιόλας από ό,τι άλλα μοντέλα. Όχι, είμαστε πολύ κοντά στις δεσμεύσει του κυρίου Λάντ κατά την προκλητική του εκστρατεία. Με ριζοσπαστικέ ε, μεταρρυθμίσει και στην αρχή των χρηματοδοτικών ε, αγορών δεν υπήρξε και αποθέωση στην στο άκουσμα των προτάσεων. Δεν ήταν όλοι πολύ ευχαριστημένοι με αυτές τις προτάσει που ακούστηκαν. Όμως άλλοι όπω εσεί φαντάζομαι θα θεωρήσουν ότι δεν πάμε αρκετά μακριά. Κάποιοι, προφανώς, εάν κάποιοι λένε ότι οι προτάσεις μας ε, δεν είναι αρκετά ριζοσπαστικές, ενώ κάποιοι πιστεύουν το αντίθετο, αυτό φαίνεται να δείχνει ότι δεν είμαστε πολύ μακριά από την αλήθεια. Δηλαδή να γίνει μια μεταρρύθμιση χωρίς όμως να βλάψουμε δομές που μέχρι τώρα έχουν αποδείξει την αποτελεσματικότητά τους. Τεσσερά λεπτά εξαιρετικά. Ε, περνάμε στην ΚΟΕ τώρα. Γιώργεν παρακαλώ. Ευχαριστώ, μια ερώτηση προς τον κύριο Σόιμπλε. Είπατε ότι η πολιτική της Τρόικα είναι, λέτε, επιτυχής. Μα πώς εξηγείτε ότι διευρύνεται η απόσταση πλούτου και φτώχειας στην Ευρώπη. Είχα πάει στην Ελλάδα και είδα να υφίστανται πιέσεις οι τράπεζες γιατί μετά την πολιτική λιτότητα ο κόσμος δεν μπορεί να αποπληρώσει τα ε, δάνειά του και τις τελευταίες εβδομάδες ή και μήνες διαβάζουμε στις ε, γερμανικές εφημερίδες ότι η λιτότητα έχει επηρεάσει και τις γερμανικές εξαγωγές. Τη βιομηχανία μας λοιπόν. Πώς θέλετε να μειώσετε αυτή την ψαλίδα ε, ε, και να καταργήσετε τη διαφορά και ποια είναι τα συγκεκριμένα εργαλεία και μέσα που θεωρείτε κατάλληλα για να δημιουργηθεί ανάπτυξη και πλούτους και για τους άλλους στην Ένωση γιατί δεδομένου ότι οι Γερμανοί και άλλες χώρες θέλουν να περικόψουν και τα γερμανικά και τα ε, γενικότερα ευρωπαϊκά κονδύλια και πώς θα ανακτηθεί και πώς θα αυξηθεί η εμπιστοσύνη των πολιτών, ανδρών και γυναικών. Γιατί πιέζονται και, και αποκλείονται όλο και περισσότερο κοινωνικά αυτοί οι άνθρωποι. Η απάντηση από την τελευταία ερώτηση ε, προκύπτει ως εξής. Προσπαθούμε να διατηρήσουμε και να εξηγήσουμε ακριβώς πώς έχουν οι συσχετισμοί. Μπορεί να διαφέρουμε στις απόψεις μας, αλλά για όλα τα προβλήματα δεν θα πρέπει να ε, κατηγορείται η Ευρωζώνη, οι κυβερνήσεις, η Ευρωπαϊκή Ένωση. Με κάποιες πολιτικές δυνάμεις στη Γερμανία έχουμε πρόβλημα και ε, αγωνιζόμαστε να εξηγούμε ε, ότι δεν θα έρθει ανάπτυξη με την αύξηση του δημοξίου χρέους. Σε όλες τις εθνικές οικονομίες όλοι οι οικονομολόγοι λένε ότι όσο περισσότερη είναι η συμμετοχή και το ποσοστό του κράτους στην οικονομία τόσο χαμηλότερη είναι η ανάπτυξη. Προσπάθησα την ε, περασμένη Παρασκευή και κατέβαλα προσπάθεια να εξηγήσω στη Γερμανική Βουλή τι αποφάσισε το Eurogroup, ότι η ελληνική εθνική οικονομία πρέπει να περάσει μια, ένα μεγάλο μετασχηματισμό αντίστοιχο με αυτό που πέρασαν πριν από 20 και πλέον ε, ε, χρόνια αυτό που τότε ονομαζόταν σύμφωνο της Βαρσοβίας τέτοια κράτη και αυτή δεν είναι απλή πρόκληση και δεν θα πρέπει να τρέφουμε αυταπάτες για αυτό το γεγονός και το άνοιγμα της ψαλίδας ε, στην κοινωνία μας ε, και φαίνεται από διάφορες στατιστικές, αλλά κατά την άποψη της γερμανικής κυβέρνησης το αίτιό της είναι ε, η επιτάχυνση των μεταρρυθμίσεων και των αλλαγών που έχουν επέλθει από την παγκοσμιοποίηση συμπεραυμανωμένων και των αλλαγών με τις σύγχρονες ε, τηλεπικοινωνίες. Κοιτάξτε, οι αγορές εργασίας πώς αλλάζουν όλο και περισσότερο υπάρχει ανταγωνισμός για θέσεις εργασίας απανταχού της γης και είναι τελείως διαφορετική η πίεση. Στον Μπαγκλαντές είδαμε τις πυρκαγιές, τη θεομηνία. Και ε, αντίστοιχα πριν από μερικές δεκαετίες έτσι, είχε καταστραφεί η ε, γερμανική κλωστοϊφαντουργία. Αυτές είναι αλλαγές παγκόσμιες και για να απαντήσεις χρειάζεται μεγάλη καινοτομία, επενδύσεις και της ε, εθνικής οικονομίας ε, σε ένα, ε, όλο ένα και πιο παγκοσμιοποιημένο κόσμο. Αλλιώς θα πρέπει να γυρίσουμε πίσω σε ένα δρόμο που τερματίστηκε το 1990 στην Ανατολική Ευρώπη. Ευχαριστώ Γιώργη, θέλει να επανέλθει. Ναι, συγκεκριμένα μέτρα όμω δεν άκουσα κύριε Σόεμπλε. Εντάξει, μακροπρόθεσμα μπορεί να ισχύουν αυτά που λέτε, αλλά τα συγκεκριμένα μέτρα που θα είναι σήμερα αποτελεσματικά και πώς θα αυξηθούν τα έσοδα, πώς θα αυξηθούν οι φόροι. Δεν απαντήσατε σε αυτό. Αγαπητέ συνάδελφε, ποια είναι η απάντηση. Για τη Γερμανία τα τελευταία τρία χρόνια έχει γίνει μια εντατική συζήτηση. Στην αρχή, όταν ε, ανέλαβα ε, τα καθήκοντά μου, τέλη του 9, αρχές του 10, ε, με επέκριναν ότι μειώναμε πολύ γρήγορα τα ελλείμματα στη Γερμανία δήθεν και περιορίζαμε την ανάπτυξη. Και ε, οι Αμερικανοί συνάδελφοί μου και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέφραζαν αυτό το φόβο. Στο μεταξύ σε όλες τις διεθνείς εκθέσεις και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής φερόμαστε να ε, τηρούμε όλες τις προϋποθέσεις και τις υποχρεώσεις. Και αυτό δεν ισχύει για τα κράτη-μέλη. Και εκθέσεις ε, του ΟΟΣΑ και του Διεθνούς Χρηματοοικονομικού Ινστιτούτου έχουμε αυξήσει την εσωτερική ζήτηση γιατί ανακτήσαμε την εμπιστοσύνη. Και η πιο πρόσφατη έκθεση του ΩΣΑ λέει ότι ε, το βασικό πρόβλημα για την ανάπτυξη είναι ότι αυξάνεται η κρίση εμπιστοσύνη, η δυσπιστία. Αυτοί οι προπολογισμοί ε, και αυτά τα χρέη δεν είναι βιώσιμα ε, και γι' αυτό ο κόσμος δυσπιστεί και δεν τονώνεται η ζήτηση. Και είπε και ο Αμερικανός Υπουργός ε, οικονομία ότι θα προσανατολίσει την αμερικανική οικονομική πολιτική στη γερμανική. Θα την κάνει, λέει, more German-like. Ε, το ΕΛΚ και ο, κύριος Λάγκεν. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω πάρα πολύ ε, για τα όσα μας είπατε και ο κύριος Μπαρνιέ είπε ότι το δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε στο αγώνα που δίνει η Ευρωζώνη κατά των αγορών. Η ομάδα της Ευρωζώνης πρέπει να αλλάξει προπονητή. Ε, αναρωτιόμαστε, είπε ο κύριος Σόιμπλε πριν τα προβλήματα και με την Κεντρική Τράπεζα. Ο κύριος Μοσκοβισή ε, θέλει να αλλάξει ε, γήπεδο. Ε, ε, θέλω να ρωτήσω και τους δύο υπουργούς, και τον Γάλλο Υπουργό, Είπατε ότι θέλετε δημοκρατικό έλεγχο στην Ευρωζώνη, κοινό όριο για το χρέος και τα λοιπά και αυτό χρειάζεται αναθεώρηση των συνθήκων. Πότε βλέπετε να υπάρχει ρεαλιστικά τέτοια ευκαιρία. Και μια ερώτηση προς τον Γερμανό Υπουργό Οικονομικών. Είπατε ότι πρέπει να λυθούν ορισμένα νομικά ζητήματα για την Τραπεζική Ένωση, ιδιαίτερα σε ό,τι έχει να κάνει με τη συμμετοχή των μη μελών της Ευρωζώνης και την ανεξαρτησία της ΕΚΤ, αλλά και τη συμπερίληψη όλων και ε, του κειμένου της συνθήκης στο 27 εδάφιο 6 προβλέπει αυτή περιορισμούς. Πώς θα το λύσετε αυτό και πού υπάρχουν δυνατότητες ακριβώς επίλυσης. Ευχαριστώ. Oui, je crois beaucoup euh, ναι, πραγματικά πιστεύω και εγώ ότι χρειάζεται ενισχυμένο δημοκρατικός έλεγχος ε, στη ζώνη ευρώ ε, πριν από πολύ καιρό, όταν ήμουν νέο, ήμουν υπουργό οικονομικών και πήγαινα σε διάφορα συμβούλια, μεταξύ των οποίων και το Συμβούλιο Εξωτερικών. Ήμουν εδώ, ήμουν στη συντακτική συνέλευση. 15 χρόνια από τη ζωή μου πέρασα στα θεσμικά όργανα. Και επανερχόμενο στο ΕΚΟΦΗΝ, ε, βλέπω την Ευρώπη και δεν έχω την αίσθηση ότι βελτιώθηκε ο μηχανισμός λήψης αποφάσεων. Το αντίθετο, είναι όλα πιο περίπλοκο, είμαστε πολυάριθμοι, είμαστε, είναι ετερογενής πλέον η Ευρωπαϊκή Ένωση, περισσότερο από το παρελθόν, ε, ακολουθούνται διαφορετικές τεχνικές, δεν λειτουργεί το σύστημα. Το Eurogroup έχει φοβερή ισχύ. Αυτός ο θεσμό το συζητούσαμε με τον κύριο Ντράγκη, είναι το πιο λειτουργικό κομμάτι τη Ένωση. αλλά ειλικρινά δεν έχουμε μηχανισμούς ε, που αντιστοιχούν αναλογικά στην ισχύ αυτού του θεσμού. Είδατε πόσε μέρε χρειάστηκαν για να πάρουμε την απόφασή μα και γι' αυτό σα είπα ότι εν τέλει αυτό πρέπει να γίνει στην Ευρωζώνη και γι' αυτό πιστεύω ότι ε, πρέπει να γίνει σεβαστή η ακαιρεότητα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ναι, μεν, αλλά θα πρέπει να βρει τον τρόπο με τον οποίο θα νομοθετεί, θα ελέγχει, θα παρακολουθεί πιο αποτελεσματικά για να υπάρχει στενότερη σχέση ανάμεσα στα θεσμικά όργανα. Ε, μάλλον θα χρειαστεί η τροποποίηση των συνθήκων και αυτή είναι η προσωπική μου άποψη. Η άποψη ενό Ευρωπαίου αλλά και του Υπουργού Οικονομικών. Δεν είμαι κατά τη τροποποίηση ε, των συνθήκων, αλλά πραγματικά δεν πιστεύω ότι είναι το πλέον επίγον ζήτημα. Υπάρχουν άλλα που είναι πιο επίγοντα. Ε, σε κάθε περίπτωση ε, ε, έχουμε τις ευρωπαϊκές εκλογές το 2014. Αυτό έχει πολύ μεγαλύτερη σημασία. Αλλά ως πολίτης και πάλι σας λέω αυτό το θέμα της αλληλέγγυας ενσωμάτωσης, της σχέσης ανάμεσα της εμβάθυνσης της ζώνης ευρώ και του δημοκρατικού ελέγχου είναι στοιχεία που πρέπει να προκύπτουν όλο, στο δημόσιο διάλογο με όλους τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στη συνέχεια είμαι ανοιχτό σας, κάνουμε και ντροπή των συνθήκων, αλλά υπάρχουν άλλα πιο επίγοντα. Ευχαριστώ. Για ε, αγαπητέ συνάδελφε Λάγκεν, στην περασμένη συνεδρίαση του ΕΚΟΦΗΝ παρακαλέσαμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τις νομικές υπηρεσίες να μελετήσουν πώς μπορεί κανείς με περιορισμένη τροποποίηση των συνθηκών να λύσει το πρόβλημα. Σύμφωνα με το άρθρο 127.6 για την ερμηνεία από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ε, είναι δύσκολο να λυθεί ε, και το είπατε και εσείς ο ίδιος. Ε, ο Σουηδός συνάδελφος που έκανε αυτή την πρόταση και την παράκληση πρόσθεσε ότι αν μπορούσαμε να συμφωνήσουμε να ακολουθήσουμε αυτό το δρόμο μπορούμε να βρούμε και μία ενδιάμεση λύση. Περιμένω το αποτέλεσμα στην αυριανή συνεδρίαση, δυστυχώς ακόμα δεν το έχω λάβει εκ των προτέρων. Are you happy with that, Σε ικανοποιεί αυτή η απάντηση, Βέρνερ. Ναι. Έχω και άλλη ερώτηση όμως προς τον Γάλλο Υπουργό. Ε, το ο κοινό ε, όριο ή ο περιορισμός του χρέους. Εδώ πέρα ε, μπορείτε να συμπεριλάβετε και τα ευρωομόλογα. Ναι, η Γαλλία καταρχήν θα ήταν υπέρ τη έκπτωση των ευρωομόλογων Αυτό το είπαμε και στην προεκλογική μα εκστρατεία και στα Ευρωπαϊκά Συμβούλια. Το έχουμε συζητήσει και με του εταίρου μα. Κύριο Σόιμπλε, μα είπε βέβαια ότι αυτό αποτελεί χωριστικό όριο. Όμως να μην ξεχνάμε ότι στο τέλος της όλης διαδικασίας θα μπορούσε να είναι αυτό μια λύση. Θα μπορούσε να είναι το όριο, το... η απόλυξη. Πριν όλα τα υπόλοιπα ενισχυθούν όπως τα εξηγήσαμε με την αλληλεγγύη και την ολοκλήρωση, την πολιτική και την ε, εξηγήση του χρέους, αυτά θα μπορούσαν να ακολουθήσουν. Για τους σοσιαλιστές, ε, πείτε Σιμών, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αποφάσισε την τραπεζική εποπτεία ως προϋπόθεση για την ανακεφαλαιοποίηση. Ως όρο. Αλλά σε αυτή την πρόταση λέει ως έναν όρο. Και αυτό αποκτά νέα σημασία σύμφωνα με αυτά που μας λέει και ο κύριος Σόιμπλε. Δεν είναι ο μοναδικός όρος, είναι ένας όρος. Αλλά εμείς στο Κοινοβούλιο θεωρούμε άμεση ε, ανεκεφαλαιοποίηση από τον ESM σκόπιμη. Και θα πρέπει να τονίσουμε όμως ότι ε, παραμένουν αυτά χρήματα των φορολογουμένων και από τον ESM. Τα μοναδικά κονδύλια και τα μοναδικά ταμεία που μπορούμε εμείς να συλλέξουμε στην Ευρώπη που εφαρμόζουν αυτά που έχουμε υποσχεθεί στον κόσμο, δηλαδή να μην επιβαρύνουμε στο μέλλον το φορολογούμενο, αλλά τις ίδιες τις τράπεζες είναι ε, ένα ταμείο εγγύησης των καταθέσεων και ένα ταμείο ε, αναδιάρθρωσης. Το ταμείο εγγύησης των καταθέσεων το θεωρούμε ε, εμείς προτιμότερο και σωστό, όπως και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τουλάχιστον, αν καταρρεύσει μια μεσαία τράπεζα, δεν θα επιβαρυνθεί έτσι ο φορολογούμενος σε κάθε κράτος μέλος. Ε, το έχουμε αποφασίσει εδώ και καιρό ε, στο ε, Κοινοβούλιο και περιμένουμε το Συμβούλιο να δεήσει να συμφωνήσει. Εδώ και μήνες δεν κινείται τίποτα. Το δεύτερο ταμείο ανακεφαλαιοποίησης έχει ένα ποσό που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρεί ότι μπορεί να επιβληθεί πολιτικά στο Συμβούλιο. 1,0% των καταθέσεων. Βλέπε 77 δισεκατομμύρια ευρώ. Αν κοιτάξουμε όμως η κρίση μέχρι τώρα, τι απαιτεί ως μέτρα ανακεφαλαιοποίησης, αναδιάθρωσης για τις τράπεζες, μας βγαίνει το διπλάσιο και πλέον. Πέρα από τα άλλα εργαλεία, το bailing και τα λοιπά που προβλέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, είναι πολύ χαμηλό αυτό το ποσό. Και σας ερωτώ και εδώ, εάν θέλουμε να τηρήσουμε τις υποσχέσεις μας το φορολογούμενο ότι στο μέλλον θα τον κρατήσουμε μακριά από τους κινδύνους σε ό,τι αφορά το ποσό αλλά και τη δέσμευσή σας ότι επιτέλους ε, θα ξεφύγουμε από αυτό και θα ολοκληρώσουμε την νομοθεσία ιδιαίτερα για την εγγύηση των καταθέσεων. Τι θα κάνουμε έτσι ώστε να μην επιβαρύνεται ο ESM και τελικά τα χρήματα των φορολογουμένων να μην είναι το μοναδικό μέσο που έχουμε στα χέρια μας. Αυτό βασικά ήταν για σένα γκολφ. Όχι, όχι και προς τους δύο. Ένα λεπτό έκαστος τότε για να απαντήσει. Κύριο Σόιμπλε. Καταρχάς, θα πρέπει να πούμε στον κύριο Σίμων τα εξής. Όσα μέτρα και αν παίρνουμε, θα πρέπει πάντα να φροντίζουμε η χρήματα αγορά, ο χρηματοοικονομικός τομέας να μην ε, αποδυναμώνεται. Το είδαμε και με την τραπεζική κρίση. Και ο προκάτοχος μου, ο κύριος Στάιμπροκ, το αντιμετώπισε αυτό ναι, ναι, ναι, ο κύριο Στάιμπροκ ήταν τότε, θυμάστε, υπουργό Οικονομικών. Τώρα στη Γερμανική Βουλή έχει άλλα καθήκοντα αυτόν τον καιρό, αλλά βγάλαμε τα διδάγματά μας. Και στη βασιλεία 3 γιατί είναι και παγκόσμια τα θέματα. Θα πρέπει να βλέπουμε την ανταγωνιστικότητά μας στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα διεθνώς και παγκοσμίω. Γιατί η λειτουργικότητα των τραπεζών έχουν να κάνουν με ανάπτυξη, με απασχόληση. Έχουμε τη διαδικασία ε, Βασιλείας 3. Ε, Ελπίζω ε, πλέον η οδηγία ε, για ε, τις κεφαλαιακές απαιτήσει 4, CDR 4 επιτέλου, να λυθεί φέτο και ε, απευθύνω έκκληση και προς εμάς, δεν είναι το θέμα και το πρόβλημα στο Συμβούλιο. Στη συνέχεια, θα πρέπει να δούμε τι γίνεται και στις τράπεζες. Υπάρχει το CDR4 ε, και η Βασιλεία 3, αλλά και στη Γερμανία ε, ιδρύσαμε ένα εθνικό ταμείο ανασυγκρότησης. Αλλά ε, για την ε, εγγύηση των καταθέσεων έχουμε εθνικά συστήματα ο καθένας διαφορετικά. Αν αυτό τον καιρό με τα παρόντα δεδομένα ε, θέλετε να εξοευρωπαίσετε τα συστήματα ή να κάνετε κάποια μεταβατικά συστήματα μεταξύ των διαφόρων εθνικών συστημάτων εγγύησης καταθέσεων Μην έρχεστε και ρωτάτε πώς θα εγγυηθούμε τη συμφωνία των πολιτών μας απέναντι σε ευρωπαϊκά ζητήματα. Θα είναι πάρα πολύ ισχυρή η αντίσταση. Δεν θα έπρεπε να ακούσουμε απάντηση από τον κύριο Μοσκοβίτση γιατί εξέπνευσε ο χρόνος. Ε, θέλετε απάντηση, αλλά θα στερήσετε μια ερώτηση από έναν συνάδελφο. Μια σύντομη απάντηση, παρακαλώ. Να να απαντήσω πολύ γρήγορα. Σε ό,τι μας αφορά, έχουμε κάνει σχετισμό μεταξύ της ε, τραπεζικής εποπτείας τις εξηγήσεις των τραπεζών. Εδώ θα πρέπει ο μηχανισμός αυτός να είναι ένα μέσο στήριξη. Όμω για μένα η Τραπεζική Ένωση δεν σημαίνει απλώ την τραπεζική εποπτεία. Μιλάμε για ένα τρίπτυχο. Το οποίο θα πρέπει να ασχοληθεί και με την εγγύηση των καταθέσεων και την επίλυση του θέματο αυτό. Στο, κονσέγιο, στο Συμβούλιο ε, επικεντρώνονται περισσότερο στην εποπτεία. Εμείς πρέπει να δούμε και το άλλο σκέλος. Ε, Ωραία, προχωρούμε τώρα Ευχαριστώ, Σάρον. Θα απευθύνομαι στον Υπουργό Σόιμπλε. Ε, τα κράτη εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης που μετέχουν στον ενίο μηχανισμό εποπτείας. Ε, τροποποιήθηκε σε μεγάλο βαθμό η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ούτως ώστε τα κράτη που δεν ανήκουν στην Ευρωζώνη αλλά παρόλα αυτά θέλουν να μετάσχουν στο σύστημα να μην έχουν προβλήματα. Όμως ε, στο Κοινοβούλιο δεν λύσαμε το θέμα ε, του δημοσιονομικού τέλματος, fiscal backstop, γιατί θα υπάρξουν δημοσιονομικές επιπτώσεις για αυτά τα κράτη. Οπότε μία, ένα αλλακτικό σενάριο είναι να ανοίξουμε την ανακεφαλοποίηση των τραπεζών και στα υπόλοιπα κράτη εκτός Ευρωζώνης, αλλά φυσικά θα συνεισφέρουν στο μηχανισμό αυτά τα κράτη, όμως αυτό προϋποθέτει τροποποίηση της συνθήκης. Δεύτερο εναλλακτικό σενάριο ε, μια πρόταση που τώρα τροποποιείται ε, να δούμε το κομμάτι του EFSM διευκόλυνση ε, του ισοζυγίου τρεχουσών πληρωμών για κράτη εκτός ευρωζώνης αλλά αυτό διαφοροποιείται από την παρέμβαση της ανακεφαλαιοποίησης τράπεζας δεν εντάσσεται στο ισοζύγιο τρεχουσών πληρωμών λοιπόν το δημοσιονομικό πρόβλημα αυτών των κρατών που θέλουν να μετάσχουν στο μηχανισμό αλλά δεν ανήκουν στην ευρωζώνη πώς αντιλαμβάνεστε εσείς. Καταρχάς κυρία Χιούπνερ, θα ήθελα να ξανατονίσω ότι βέβαια δεν μας αρέσει να τα ακούμε πάντα, αλλά ισχύει αυτό. τραπεζική εποπτεία δεν δημιουργεί ακόμα κατάσταση όπου κάθε τράπεζα μπορεί να ανακεφαλαιοποιείται άμεσα από τον ESM θα χρειάζεται ως προϋπόθεση ακόμα αίτηση κράτους μέλους και εφαρμογή προγράμματος προσαρμογής. Αυτή είναι η αιρεσιμότητα. Δεν, δεν καταργείται του μηχανισμού ε, σταθερότητας. Οπότε τα κράτη που δεν συμμετέχουν στην Ευρωζώνη ε, έχουμε το πρόβλημα πραγματικά να υπάρξει ίση μεταχείριση. Το είπα και στην αρχή οι μετά οι χώρες που δεν συμμετέχουν στο ευρώ θα πρέπει να κληθούν να αποφασίσουν τι επιθυμούν. Αν είναι πραγματικά ένα τμήμα του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Προστασίας ή με ποιο τρόπο. Η δική μου φαντασία δεν επαρκεί για να φανταστεί πώς ένα κράτος μπορεί να μπει στο μηχανισμό στήριξης χωρίς να είναι μέλος της Ευρωζώνης. Δεν ξέρω αν βρούμε κάποιο άλλο τρόπο, αλλά επαναλαμβάνω, ε, ο μηχανισμός του, της ε, σταθερότητας ποιος είναι. Πάντα ένα κράτος μέλος έρχεται και υποβάλλει αίτηση να ενταχθεί εκεί και υπογράφεται μνημόνιο, συμφωνείται μνημόνιο. Σε καμία περίπτωση δεν σημαίνει αυτό άμεση ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών. Did you want to come back on that, Danuta? Danuta, Υπουργέ. Όχι. Εν τη αυτή περιπτώσει η επόμενη ερώτηση από πλευράς του ΕΛΚ Τζιόγκο Φέιο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ Σάρων. Μία ερώτηση και για τους δύο υπουργού και γι' αυτό θα είμαι σύντομος. Όπως ξέρετε, πρόσφατα άλλαξαν οι όρια για τη δανειοδότηση της Ελλάδας. Στο βαθμό που θα υπάρξει και συνάντηση του Eurogroup τώρα, ήθελα να ξέρω κατά πόσον ως προς τα επιτόκια, ως προς τον, ε, τη διάρκεια του χρέους, κατά πόσον τέτοιοι όροι θα μπορούσαν να προβλεφθούν και για, τέτοια, και για άλλα κράτη που, για τα οποία ισχύουν προγράμματα της Τρόικας, όπως συγκεκριμένα για την Πορτογαλία. Δεν θα συμβούλευα την Πορτογαλία να κάνει ένα τέτοιο βήμα, διότι ε, αν ήμουν άλλο κράτος μέλος θα δίσταζα να κάνω σύγκριση με την Ελλάδα. Η Ελλάδα είναι τελείως ξεχωριστή περίπτωση, ιδιάζουσα. Γι' αυτό ε, ε, τα έχω ακούσει αυτά και από την Ιρλανδία και την Πορτογαλία. Στη συνέχεια, μειώσαμε τα επιτόκια για τα διμερεί ε, δάνεια με την Ελλάδα. Για ε, την Ιρλανδία και την Πορτογαλία δεν έχουμε διμερεί δάνεια και τέτοια προγράμματα και δεν μπορεί να μεταφερθεί αυτό. Και στο FSF προβλέψαμε ε, ε, δεκαετή ε, αναβολή καταβολής των δόσεων με επιμήκυνση του προγράμματος. Γιατί η Πορτογαλία και την Ελλανδία που έχουν πάρει το δρόμο των αγορών θα ήταν ολέθριο ένα τέτοιο σημάδι και πραγματικά θα σας συμβούλευα να μην ακολουθήσετε αυτή την ατραπό Euh, θα ήθελα να ακολουθήσω ακριβώς την ίδια κατεύθυνση. Για την Ελλάδα πρώτα απ' όλα για... χαίρομαι, αναφέρθηκα στο ότι είναι καμπή η σημερινή χρονική στιγμή γιατί θα δοθεί μια λύση σε αυτά τα προβλήματα που γνωρίζει η χώρα διατηρώντας και διαφυλάστα την ακαιρεότητα της Ευρωζώνης. Για μένα αυτό συνιστά σημαντικότατο στόχο. Τώρα για την ίδια τη συμφωνία είναι σταθερή, βιώσιμη, πλήρης και επιπροσθέτως έχουν αναλυφθεί οι δεσμεύσεις και για το μέλλον, οπότε την περασμένη εβδομάδα ζήσαμε μια ιστορική στιγμή. Έπρεπε να γίνει, ήταν επαχθής η διαδικασία και χρονοβόρα, αλλά μην ξεχνάμε πόσο περίπλοκα είναι τα ζητήματα. Τα, το σημείο εκκίνηση για όλε τι χώρε ήταν διαφορετικό, αλλά ήταν υψηλέ και οι απαιτήσει. Για να είναι σταθερό και βιώσιμο όμω το πρόγραμμα, έπρεπε να εξασφαλίσουμε και τη χρηματοδότηση του εν λόγω ε, προγράμματο και τη βιωσιμότητα του χρέου μέχρι το 2020 και μετά. Ε, είμαι σχετικά αισιόδοξο ε, ότι μετά την ε, επιτυχή επαναγορά του χρέους, αυτό ευελπιστώ τουλάχιστον και θεωρώ ότι είναι απολύτως εφικτό, θα έχουμε τον ακρογωνίο λίθο του όλου εγχειρήματο και θα κερδίσουμε χρόνο. Ουσιαστικά οι δε Έλληνε φίλοι μα θα έχουν χρόνο για να λύσουν αυτά τα μεγάλα προβλήματα. Για την Πορτογαλία και για την Ιρλανδία, όπω και ο κύριο Σόιμπλε, θα δώσω την ίδια απάντηση. Δεν είναι συγκρίσιμε οι καταστάσει και εξυπακούεται ότι δεν είναι ευκταίο να μιμηθούμε τι λύσει που ευρέθησαν για την Ελλάδα. Το αντίθετο, στην Πορτογαλία το πρόγραμμα ε, προχωρά όπως είχε προγραμματιστεί ε, ε, και ε, προσεχώς θα επανέλθει η χώρα στις αγορές. Αυτό πρέπει να επιδιώξει η χώρα σας και μπορεί να το κάνει. Θέλετε συμπληρωματική ερώτηση. Ναι. Κοιτάξτε, εγώ στηρίζω την κυβέρνηση που αυτή τη στιγμή κάνει σοβαρέ προσπάθειε στην Πορτογαλία για να εκπληρώσει τι δεσμεύσει τη. Τι κίνητρο θα δώσετε σε κράτη όπω Πορτογαλία. αναγνωρίζω στην κυβέρνηση αυτή τι προσπαθίε που κάνει και το πρόγραμμα που προσπαθεί να υλοποιήσει και μπορούμε να προσφέρουμε την πλήρη στήριξή μα ως συνήθως συμφωνώ απολύτως με τον Πιέρ Μοσκοβισή. Συνεχίστε αυτή την αγαστή συνεργασία, αλλά ξέρετε για το θέμα της βιωσιμότητας των επιτοκίων και το, του χρέους, ε, καταλαβαίνω γιατί ανησυχούν όλοι. Λίαν Βανκόκ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Για τους ε, ειδικού ε, εδώ σε αυτή την αίθουσα, ξέρουμε ότι πολλοί είναι υπέρ του φεντεραλισμού. Το επόμενο στάδιο της ευρωπαϊκής οικοδόμησης είναι η δημοσιονομική πειθαρχία στα κράτη-μέλη, αλλά και η οικονομική, το, οικονομικό το δημοσιονομικό δυναμικό, το δυναμικό του προπολογισμού σε επίπεδο ευρωπαϊκό. Και αν διαβάσουμε τι προτάσει του κ. Φανρόμποη στο ενδιάμεσο, στο ενδιάμεσο φύλλο πορείας, το blueprint, το αποτύπωμα που εξαντλούσε η Επιτροπή, την έκθεση της Station που ενέκρινε το Κοινοβούλιο πρόσφατα, χρειάζεται δυναμικό προϋπολογισμού για να αντιμετωπιστούν τα ασυμμετρικά πλήγματα και όπως είπε προηγουμένως ο κύριος Μοσκοβισή να καταρτιστούν πολιτικές αντικυκλικές για να αντιμετωπίζουν τα κυκλικά φαινόμενα. Βεβαίω το θέμα είναι πώ θα χρησιμοποιηθεί αυτό το επιπλέον δυναμικό του προπολογισμού, δηλαδή πώ θα αντιμετωπιστούν τα φαινόμενα αυτά τα κυκλικά. Όμω το πρόβλημα ουσία που για πολλού εμά εδώ το Κοινοβούλιο είναι σημαντικό και προσφυλέ είναι πώ θα τροφοδοτήσουμε αυτό το δυναμικό του προπολογισμού. Ξέρουμε όλοι εδώ ότι οι διαπραγματεύσεις για τις δημοσιονομικές προοπτικές είναι δυσχερέστατες. Πολλά κράτη θέλουν ε, να αποφύγουν την αύξηση της συνεισφοράς τους. Το ερώτημα απευθύνεται και στους δυο σας. Απλώς ο Γάλλος Υπουργός ε, πίντησε εν μέρη στην αρχική του παρέμβαση, γι' αυτό απευθύνουμε κυρίως στον κύριο Σόμπλε. Πώς μπορούμε να ενισχύσουμε πλέον τους ίδιους πόρους της Ένωσης για να μπορέσουμε να έχουμε αυτό το δυναμικό στον προπολογισμό. Τι εργαλείο, ε, δάνεια, ε, φόρους θα επιβάλλουμε. Εάν θέλουμε να ξεφύγουμε από τη συλλογιστική ε, και από του υπολογισμού αυτού που καθένα συνεισφέρει και το τι θα περιμένει να πάρει ως αντάλλαγμα. Das ist αυτό το ερώτημα δεν μπορεί να το απαντήσει κανείς έτσι με δύο φράσεις απλά. Διότι καταρχήν και επί της ουσίας και η γερμανική κυβέρνηση και ο υποφαινόμενος συμφωνούμε με την προσέγγισή σας. Πλην όμως αυτό θα απαιτεί αναθεώρηση συνθήκων. Ήδη οι πόρια απαιτούν ε, ε, ίδιους φόρους, άρα και αλλαγή συνδικών. Και για την Ευρωζώνη πώς θα ε, ρυθμιστεί αυτό και πώς θα ρυθμιστεί σε επίπεδο 27 ως θεσμικό όργανο. Εγώ είχα προτείνει να ενισχυθεί ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και σε ζητήματα που δεν αφορούν και τους 27 να αποφασίζουν οι βουλευτές που προέρχονται από τις χώρες ε, που ε, ενέχονται. Γιατί πώς μπορούμε να αποφασίσουμε για ένα προϋπολογισμό των 17 μόνο όλοι αλλά οι στοδίνεκες δεν μπορούν να τα χρηματοδοτούν όλα αυτά αποκλειστικά τα κράτη-μέλη. Δεν θεωρώ ότι θα τελεσφορήσει αυτή η προσπάθεια. Και για τον επόμενο προϋπολογισμό αλλά και για το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο θα πρέπει να προσέξουμε πάρα πολύ να μην υποτιμήσουμε το ζήτημα και την προβληματική του ηθικού κινδύνου. αν δεν διατηρηθεί η πίεση για φιδωλή διαχείριση των πόρων σε όλα τα επίπεδα, δεν πρόκειται να πείσουμε τους ευρωπαϊκούς λαούς για την ευρωπαϊκή αυτή πορεία. Χρειάζεται προσοχή και το έδειξαν αυτό και οι διαπραγματεύσεις ε, τη περασμένη εβδομάδα στο Συμβούλιο. Ε, Όπως είπε ο απέντησα εν μέρη στην προκαταρκτική ε, μου παρέμβαση. Απλώς να πω εδώ ότι θα ήθελα να υπάρχει ο απολογισμό για την Ευρωζώνη που θα μπορούσε να λειτουργεί για να αντιμετωπίσει και τα κυκλικά φαινόμενα με ίδιου πόρου ενδεχομένω. Υπάρχουν και άλλε ιδέε. Ο φόρο για τι χρηματοπιστικές συναλλαγές λόγου χάρη μέσω τη ενισχυμένη συνεργασία με τη συμμετοχή τουλάχιστον 11 κρατών μελών ή ο Εταιρικό φόρο για τις επιχειρήσεις. Συμμερίζουμε πάντω αυτά που λέει και ο Βόλφκανγκ για τον συγκεκριμένο δημοκρατικό έλεγχο στην Ευρωζώνη. Δεν λέω να δημιουργηθεί ένα νέο Ευρωκοινοβούλιο. Απλώ το Ευρωκοινοβούλιο όπω λειτουργεί να ενισχύσει τι αμμοδιότητέ του. σω με μια επιτροπή ε, εντεταλμένη να συζητήσει το θέμα αυτό στο 2014. Το Ευρωκοινοβούλιο είναι ένα από τα ε, σώματα που ασχολούνται ακριβώ με τα προβλήματα τη Ευρωζώνης, όπω το Συμβούλιο και το Eurogroup. Πολύ συχνά συμπεριλαμβάνονται στην μέσα διάταξη τα προβλήματα τη Ευρωζώνης. Um, Η τελευταία ερώτηση, Γκούναρ Χόκμαρκ από το ΕΛΚΑ. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους υπουργούς γιατί τη σημερινή τους παρουσία τα όλα ζητήματα της ανταγωνιστικότητας και της σταθερότητας εγγράφονται στη συζήτηση της Ευρωζώνης ή όχι, τα συν και τα πλήν ε, υπάρχουν πάντοτε και ε, εγώ προσωπικά ανησυχώ πάρα πολύ διότι το στένος Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι η ίδια Ευρωπαϊκή Ένωση και υπάρχει κίνδυνος ε, κατακαιρματισμού των αγορών των χρηματοπιστωτικών αγορών, αλλά όχι μόνο και του εποπτικού μηχανισμού. Θα ήθελα λοιπόν οι Υπουργοί να μου πούν πώς αντιλαμβάνονται την ύπαρξη αυτή των, αυτών των κινδύνων και των επιπτώσεών τους. Μήπως θα έπρεπε να εισηγηθούμε τροποποίηση των συνθήκων για να μπορέσουν να μετάσχουν όλοι στις μελλοντικές δομές. Δεύτερον, για την ανταγωνιστικότητα, εφόσον μιλάμε για opt-in και opt-out ε, για διάφορα θεσμικά συστήματα, τι γίνεται σήμερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ε, τι χρειάζεται ε, ούτως ώστε οι κυβερνήσεις να μπορέσουν να προωθήσουν τι ε, τις ε, μεταρρυθμίσεις που σχετίζονται με την ανταγωνιστικότητα και να επιτύχουν σταθερότητα σήμερα. Στρέφομαι προς τον ε, Υπουργό Μοσκοβίτση. Υπάρχουν κάποιοι συγκεκριμένοι θεσμοί που χρειαζόμαστε, παραδείγματο χάρη. Μήπως χρειαζόμαστε για τις κρατικές ενισχύσεις και την εθνικοποίηση των χαλιβουργιών. μήπω λέω, χρειάζονται νέοι κανόνε, Wolfgang, νομίζω ότι θα έπρεπε εσύ πρώτα να απαντήσει ή να το αφήσουμε στον Πιέρ. Ο Πιέρ θα, απαντήσει, θα αποφασίσει ποιος θα απαντήσει πρώτος. Για την Χαλιβουργία έχει δοθεί ήδη απάντηση. Δεν ήταν η λύση που είναι η γαλλική κυβέρνηση. Το ξέρετε. Είναι ένα αποτρεπτικό μέσο. Και τα αποτρεπτικά μέσα έχουν φτιαχτεί για να μην χρησιμοποιούνται εκτός σε περιπτώσεις ε, απόλυτης ανάγκης, σπάνιες, όπως η χρήση των πυρηνικών όπλων. Πάντως, η ιδέα ότι η προσωρινή εθνικοποίηση ήταν κάτι το πιθανό ήταν χρήσιμη. Έχει γίνει αυτό και στις ΗΠΑ. Γι' αυτό πάντως και το αποτέλεσμα της συζήτησης ήταν τέτοιο στην ε, όλη η με τον κύριο Μιτάλη τώρα βεβαίω τον ειδικό χαρακτήρα τη Ευρωζώνη θέλουμε να τον διατηρήσουμε. Αυτό προσπαθούμε να κάνουμε και με την Τραπεζική Ένωση και ε, στο ΕΚΟΦΗΝ, αύριο θα συζητήσουμε το θέμα αυτό. Πρέπει η εποπτεία να βρίσκεται υπό τον έλεγχο τη Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα με εθνικού επόπτε. Θα πρέπει το κύρο τη τράπεζα αυτή να γίνεται σεβαστό και τα κράτη που βρίσκονται εκτό Ευρωζώνη, όταν μιλάμε για εσωτερική αγορά, να αισθάνονται ότι η ώρα του παιχνιδιού είναι ισότιμη. Θα καταφέρουμε λοιπόν έτσι το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα. Πιστεύω ότι η Ευρωζώνη μπορεί να ξεπεράσει τα όρια της ενισχυμένης συνεργασίας. Είναι συνεργασία επί της ουσίας. Αλλά η Ένωση είναι μια Ένωση των 27. Δεν είναι ομάδες των ΜΕΝ και των ΔΕ. Και αυτό ακριβώς επιδιώκουμε να ενισχύσουμε. Κύριε συνάδελφε Χέκμαρκ, προηγουμένως σε μια άλλη απάντηση είπα ότι είμαι πολύ προσιλωμένος στην υπόθεση της ίσης μεταχείρισης των κρατών μελών της Ευρωζώνης και των μη ε, μελών της Ευρωζώνης σε περίπτωση ενιαίας τραπεζικής εποπτείας. Δεν χρειάζεται να το επαναλάβω. Θα πρέπει να βρούμε μια αρρύθμιση. Αυτό είναι απαραίτητη. Να προσθέσω ακόμα ότι αν δεν θέλουμε να έχουμε εμβάθυνση των διαφορών και μεγαλύτερη απόσταση των 17 και των 10, θα πρέπει οι 10 να συμμετέχουν όσο γίνεται. Θα ήταν χρήσιμο να λένε και οι 10 ή όχι όλοι ενδεχομένω, αλλά όσο γίνεται περισσότεροι να δηλώσουν ότι θέλουν να συμμετέχουν στην εποπτεία ή να δούμε βλέποντας και κάνοντας για να δούμε πώς θα περπατήσει και μετά να συμμετέχουμε. Θα ήταν χρήσιμο όσο γίνεται περισσότεροι από τους 10 να δηλώσουν συμμετοχή. Και επίση αν θέλουμε να ενισχύσουμε την Ευρώπη και για μια υφόρο και βιώσιμη ανάπτυξη στην παγκόσμια οικονομία, οφείλουμε στην Ευρώπη να επιλέξουμε περισσότερο και ισχυρότερο το δρόμο και της πολιτικής ε, ολοκλήρωσης. Γι' αυτό και η ΟΝΕ, που είναι και τμήμα των συνθηκών, Δηλαδή όταν κάποιο στηρεί τις προϋποθέσεις οφείλει να γίνει μέλος της ΟΝΕ, δεν θα πρέπει να παραγνωρίζεται ή να παραβλέπεται. Ήταν σωστή απόφαση και αν δεν την είχαμε λάβει πριν από 10 χρόνια θα έπρεπε να τη λάβουμε επιγόντω τώρα. Γιατί όταν έχεις ένα κόσμο παγκοσμιοποιημένης οικονομίας δεν έχει καμία πιθανότητα ως Ευρωπαίος εάν δεν συνεχίσει την ολοκλήρωση. Και αν βαθύνει το χάσμα μεταξύ των 27 ε, αυτό δεν είναι ένα θέμα που επιβαρύνει κατά κύριο λόγο ότι είναι πρόκληση για τους 17, είναι πρόκληση για τους 10. Και παρακαλώ να είναι στην αιχμή του δώρατος της ολοκλήρωσης, όσο γίνεται περισσότεροι από τους 10 αυτούς. Thank uh, Σας ευχαριστούμε. Να ευχαριστήσω αμφότερους υπουργού για το χρόνο που μας διέθεσαν. Θα θέλαμε να σας κρατήσουμε και περισσότερο, αλλά γνωρίζω ότι πρέπει να αποχωρήσετε γιατί δεν μπορούμε να αναβάλουμε την έναρξη του Eurogroup παραμείνετε σας παρακαλώ στην αίθουσα γιατί υπολείπονται οι ανακοινώσεις της Προέδρου και δεν θέλω να σας πω τι γίνεται με... Δεν θέλω να κάνω ανακοινώσεις για τους τριμερείς διαλόγους ενώπιον μιας άδεια αίθουσα, αλλά δύο λεπτάκια δώστε μου να αποχαιρετήσω τους υπουργούς και επανέρχομαι. Okay. Σας ευχαριστώ πολύ. Συνάδελφοι, ησυχία λίγο. Να σας κάνω τις αναπομείνασες ανακοινώσεις για να σας ενημερώσω για την εργασία που γίνεται στους τριμερείς διαλόγους. Σας παρακαλώ, μην ε, συνεχίσετε ιδιωτικές συνομιλίες. Please. Please, I know it's all very Ξέρω ότι είναι πολύ ενδιαφέροντα αυτά, αλλά όσο πιο γρήγορα τελειώσουμε τι ανακοινώσει, τόσο πιο γρήγορα θα μπορέσουμε να συνεχίσουμε. Για την οδηγία για τι κεφαλαϊκέ απαιτήσει και το κανονισμό, πολιτικό τριμερή διάλογο είχαμε την περασμένη Πέμπτη για θέματα ρευστότητας, μόχλευση ε, και τα λοιπά και τεχνικές διαπραγματεύσεις και Δύο τριμερείς διαλόγους αναμένεται να έχουμε στο Στρασβούργο την άλλη εβδομάδα, την Τρίτη και την Πέμπτη. Για το, ε, τη δέσμη των δύο οδηγιών του ΠΑΚ, 13 Νοεμβρίου, ο, ο τριμερής διάλογος, συζητήθηκαν θέματα που εκκρεμούσαν τις εκθέσεις Γκοζές και εκθέσεις Φερέιρα για νέα διατύπωση, νέο τρόπο οικονομικού διαλόγου, ε, ρήτρα αναθεώρησης, κατεξιοδότηση πράξης, δημόσιες επενδύσεις, πώς εντάσσονται σε μεσοπρόθεσμους στόχους, δήλωση Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το λεγόμενο ε, ζήτημα του κεφαλαίου 3, ιδιαίτερα για ε, βήματα και πώς θα έχουμε ένα ταμείο εξαγοράς του χρέους. Έχουν κατατεθεί τώρα τα κείμενα και ε, η πρόταση για τη διατύπωση Ευρωπαϊκής Επιτροπής και θα συζητηθεί και ελπίζουμε να έχουμε και σύντομα ικανοποιητική έκβαση. Και κλείνει το μικρόφωνο της Πρόεδρου. Ε, για τους οίκους αξιολόγησης ε, επιτεύχθη συμφωνία στις 27 Νοεμβρίου στο τριμερή διάλογο για ε, ζητήματα ε, αξιολόγηση, ανταγωνισμού και θα συναφεί και ελπίζουμε τον Ιανουάριο ή τον Φεβρουάριο να ψηφίσουμε στην Ολομέλεια. Εδώ ολοκληρώνονται οι ανακοινώσει, διάφορα δεν έχουμε. Επόμενη συνεδρίαση την 5η 6 του μηνό, 9 με 12.30. Ευχαριστώ πολύ. Χαίρετε.